Αν όχι, θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Αγαπητέ κυρίε και κύριοι, σα παρακαλώ, θα θέλαμε όλοι μαζί να χαιρετήσουμε τον κύριο Μιαλίσκη ε, στα θεωρία που είναι πρόεδρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κέντρου Βιέσνα, λευκορώσο συγγραφέα. Αγαπητέ κύριε Μπιαλίτσκι, στις 21 Ιουνίου μετά από τρία σχεδόν έτη φυλάκισης απελευθερωθήκατε το κοινοβούλιο αυτό σε διάφορες περιστάσεις ε, εντατικά ασχολήθηκε για την απελευθέρωσή σας και ε, ζήτησε την απελευθέρωσή σας αυτής και ευτυχώ το πέτυχε στο τέλος. Σας ε, χαιρετίζουμε λοιπόν εδώ και είχατε προταθεί και για το ε, βραβείο Ζαχάροφ για την ερτρία σκέψη αύριο και χαίρομαι ιδιαίτερω λοιπόν που έχω την τιμή μαζί με του συναδέλφου μου να σα ε, καλωσορίσω εδώ ω ελεύθερο άνθρωπο. Καλωσορίσατε λοιπόν και πάλι και εκφράζω κάθε σεβασμό για το θάρρος σας και την τόλμη σας. Το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης είναι οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα εργασίας της Ιταλικής Προεδρίας. Καλωσορίζω λοιπόν εκ βάθους καρδίας εδώ στο Κοινοβούλιο τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Ματέρο Ρέντσι. Καλωσορίσατε και σας δίνω το λόγο.